once again, once again, once again, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, ladies and gentlemen, please take a seat. Παρακαλώ. Παρακαλώ καθίστε, σε ένα λεπτό θα ξεκινήσουμε. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Συμβούλιο Κορυφής της 29ης και 30ης Οκτωβρίου σχετικά με την εντολή και τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως επίσης και του υπάτου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και την πολιτική της ασφάλειας, όπως επίσης και για τη διάθεση της νέας Επιτροπής. Είμαι ευγνώμων λοιπόν προς τον Πρωθυπουργό κ. Ρέινφελτ και τον Πρόεδρο κ. Μπαρόσο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό. Κύριε Φρέντρικ Ράινφελτ, έρχεται το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, με μεγάλη χαρά είμαι ανάμεσά σας σήμερα. Θα ήθελα να σας μεταφέρω το τι συνέβη σε ένα περίπλοκο, θα έλεγα, συμβούλιο.